Presidente. E Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα πρέπει να κάνω δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά την γραπτή δήλωση την οποία κατέθεσαν οι κύριοι κύριοι Κάστεξ, Μπραντβερκ, Μπεγιόν, Πρέιντα και Βάιγκελ σχετικά με τα προγράμματα, τα ευρωμεσογειακά προγράμματα Εράσμους και Μικελάντζελο. Έχουν συλλέξει τις απαιτούμενες υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών και γι' αυτό θα αποσταλεί επί τη βάση του 123 του κανονισμού στους τελικούς του παραλήπτες με συμπερίληψη των ονομάτων όσων έχουν υπογράψει στα πρακτικά. Πρέπει να συγχαρώ λοιπόν αυτούς που κατέθεσαν τη συγκεκριμένη επιστολή. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Πεγιών για μια σύντομη παρατήρηση. Θα ήθελα εξ ονόματος των τεσσάρων συναδέλφων να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που επέτρεψαν να ληφθεί αυτή η πρωτοβουλία. Είναι ένα σαφές μήνυμα το οποίο αποστέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους εταίρους μας του Νότο και της νεολαίας εκεί. Περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ταχύτατα προτάσεις έτσι ώστε τα προγράμματα Εράσμος και Λεωνάρντο να λειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ κύριε Πεγιόν. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη ανακοίνωση του Προεδρείου. Πρόκειται για μια διόρθωση. Σας ανακοινώνω ότι η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς με